Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της Λετωνικής Δημοκρατίας, Βάλτη Σάτλας, αγαπητέ Βάλτης Σάτλας, είναι μεγάλη η χαρά που αισθανόμαστε σήμερα, που μπορούμε για πρώτη φορά να σας καλωσορίσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα καταρχάς θερμά να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα, μάλιστα, την ημέρα κατά την οποία εορτάζουμε και την δέκατη επέτειο του κοινού μας νομίσματος, του ευρώ. Ως πρόεδρος της χώρας σας και του ε, νέου αυτού μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθατε να μας ομιλήσετε. Είναι μια πρώτη φορά λοιπόν, όπως είπα νωρίτερα, και είναι και μια πρώτη φορά που ε, ανακρούστηκε ο ευρωπαϊκός ύμνος σε πανηγυρική συνεδρίαση προς τιμήν ηγέτη ευρωπαϊκού κράτους. Εδώ, μέσα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου, ε, επί τη ευκαιρία της επισκέψεώς σας, για άλλη μια φορά να αναφερθώ στην ιστορική σημασία της διεύρυνσης το 2004 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 60 χρόνια πέρασαν για να βρει η χώρα σας το δρόμο προς την ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη για να επανενωθεί και πάλι η Ήπειρός μας. Και σήμερα ζούμε όλοι σε ειρήνη, ελευθερία, δημοκρατία. Οι πολίτες μας, άνδρες και γυναίκες, χαίρουν των προοπτικών εκείνων που οι πατέρες και οι παππούδες μας μόνο να οραματιστούν μπορούσαν. Και αισθανόμαστε τη χαρά γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα ενώπιον νέων και μεγάλων προκλήσεων. Οι πολίτες της Λετωνίας το είδαν αυτό στην πράξη με τη μεγάλη οικονομική κρίση που έπληξε και τη δική σας πατρίδα, κύριε Πρόεδρε. Επίσης, η κρίση του φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πλήττει και μάλλον αποτελεί και σωστά λόγω επιπλέον ανησυχίας για τους πολίτες της Λετωνίας. Ωστόσο, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λειτουργεί βάσει τη αρχή αλληλεγγύη μεταξύ των λαών τη, αποτελεί εγγύηση. Ακριβώ αυτή τη στιγμή τη κρίσεω βλέπουμε ότι η, κοινό, η κοινότητα τη δράση, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των θεσμικών οργάνων αποτελούν το μεγάλο μα πλεονέκτημα. Από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι κρίσει, από κοινού εργαζόμαστε, μπορούμε να προχωρήσουμε απέναντι στι δυσκολίε. Και έτσι η συνθήκη της Λισαβόνας πιστεύουμε μπορεί να αποτελέσει το μέσον για καλύτερη δυνατότητα δράση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για, μια για ένα μεγάλο όπλο στα χέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Ιούνιο εφέτος προβλέπεται να δεξαχθούν εκλογές για, την... Ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προεκλογέ στα κράτη-μέλη και από κοινού μπορούμε μέσα σε μια μεγάλη δημοκρατική και ελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσουμε με το δικαίωμα της συναπόφασης για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υλοποιήσουμε αυτή την μεγάλη επιτυχία του ευρωπαϊκού οράματος και του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Δίνοντας, εκφράζω την τη ελπίδα, οι πολίτε άνδρες και γυναίκε τη Λετωνία, όπω και όλοι οι πολίτε των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η ψήφος που μπορούν να διαθέσουν ω πολίτε, ω Ευρωπαίοι, ω συνδιαμορφωτέ αυτού του κοινού εγχειρήματο και να συμμετάσχουν σε ε, αθρώα σε αυτές τις ευρωεκλογές. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά τώρα σας καλωσορίζω και παρακαλώ να λάβετε το λόγο για να απευθυνθείτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για άλλη μια φορά σας καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αξιότιμε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα καλά του λόγια, για το καλωσόρισμα και διότι με προσκαλέσατε να μιλήσω εδώ στου ε, ερετού από του λαού τη Ευρώπη. Είναι μεγάλη μου τιμή να παρευρίσκομαι εδώ εν μέσω ημών και να μπορέσω να σα ε, μιλήσω στην ε, μητρική μου γλώσσα. Ε, η γλώσσα μας ε, την τελευταία πενταετία έχει καταστεί επίσημη γλώσσα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σήμερα που σας ε, ομιλώ, οι βουλευτές που προχωρούν από τη χώρα μου διάγουν και σύντομα θα συμπληρώσουν την πρώτη τους κοινοβουλευτική θητεία, οπότε με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να ευχαριστήσω και εκείνους για την συμβολή τους. Κυρίες και κύριοι, το 2009 είναι ένα έτος πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μου. Διότι φέτος γιορτάζουμε την πέμπτη επέτειο της ε, Λετωνίας, ε, επέτειο προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στο ΝΑΤΟ. Γιατί το να ενταχθούμε στους διεθνείς αυτούς οργανισμούς, ε, ήταν στατικός μας στόχος, αμέσως μόλις ε, αποκτήσαμε την εισαρτησία μας πάλι το 1991, οπότε είπαμε ότι είναι ξεκάθαρο στόχος και η φιλοδοξία μας να μπορέσουμε να μπούμε ε, σε αυτές τις δομές, τις ευρωατλαντικές η δε διεύνηση στη δημοκρατική οικογένεια της Ευρώπης, κάτι το οποίο έλαβε χώρα κατά την πρώτη δεκαετία του αιώνα μα ήταν ε, κάτι το οποίο σηματοδότησε τις ε, σημαντικότερες αλλαγές στην Ευρώπη από τότε που δημιουργήθηκε, γεννήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια αλλαγή πάρα πολύ σημαντική, διότι η στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκαν κάποιε χώρε οι οποίε προηγουμένω ήταν απομονωμένες από αυτήν παρά την θέλησή τους. Οπότε βέβαια και ιστορικά να ληφθεί υπόψη ότι είχαμε κοινέ αξίες ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Νοεμβρίου πέρυσι εορτάσαμε την 90η ε, επέτειο δημιουργίας του κράτους μας. Πάρα πολύ σημαντικό ορόσημο αυτό για τη χώρα μας διότι ακόμα μια φορά ε, διατρανώσαμε το ότι θέλουμε να ζούμε ελεύθερα και δημοκρατικά σαν κράτος δε πράξη διακήρυξης της ε, δημοκρατίας της χώρας μας το 1918 ανέφερε επιλέξει ότι όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτως ε, εθνοτικής προέλευσης καλούνται να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν η δε Λετωνία εγγυάται ισότητα για όλους θα είναι κράτος δικαίου, κράτος δημοκρατικό χωρίς καταστολή, χωρίς την αδικία για αυτή την διάταξη είμεθα υπερήφανη. Οπότε έτσι διατρανώσαμε το ότι έχουμε πεποίθηση ε, σε αυτές τις αρχές και αυτό 30 χρόνια πριν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Ανθρώπινων Δικαιωμάτων διότι ανέκαθεν θεωρήσαμε ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και αυτό επίσης το ε, πιστεύαμε όλα αυτά τα χρόνια που εμείς αλλά και άλλες χώρες της Ανατολική Ευρώπη είχαν ε, συνδεθεί, είχαν προσδεθεί στο άρμα κάποιας χώρας που άλλα πρέσβευε. Βεβαίως και υπήρχε ειρήνη και στην Ανατολική Ευρώπη εκείνα τα χρόνια, όμως ήταν μια ειρήνη την οποία την επέβαλαν απειλές, ε, άρματα μάχης, καταστολή. Ήταν μια βαρβαρότης, μια, ένας ολοκληρωτισμός. και σας παραπέμπω στο ντοκιμαντέρ εκείνο που λέγεται The Soviet Story. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, προβλήθηκε λοιπόν και προ... σκηνοθέτης δε ήταν κάποιος λετονός. Με την ευκαιρία αυτή τώρα βεβαίως για μια φορά να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την ε, έγγραφη δήλωση της 20ης Δευτέρας Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους με την ευκαιρία της 30ης Αυγούστου ε, ως ημέρας ε, εορτασμού της μνήμης των θυμάτων του σταλινισμού. Και έτσι όλοι δεν θα ξεχάσουμε αυτά τα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα. Τώρα θα πρέπει να δούμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. kopš Φέτος έχουμε την πέμπτη επέτειο της προσχώρησης στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε με τη σημερινή συγκυρία είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρίξουμε μια ματιά, μια αναδρομή σε αυτή την πεντετία και να δούμε τι έγινε, ε, πόσο ωφεληθήκαμε, τι πετύχαμε ως Λετωνία και ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους ε, έχουμε τάξει για τη χώρα μας πρώτα-πρώτα θελήσαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ε, βόηθησε την δημοκρατία, βοήθησε το να στεριώσουν δημοκρατικοί θεσμοί στην χώρα μας Οπότε με την προσχώρηση αποδείξαμε ότι θέλουμε το μέλλον μας να είναι προσδεδεμένο με την ε, ευρωπαϊκή ταυτότητα για τις γνωστές αξίες της κοινέ μας ε, δημοκρατία, ελευθερία, υπευθυνότητα, ε, κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα και αν όχι ανεκτικότητα και ταυτόχρονα οικονομική ευημερία. Επίσης, η προσχώρηση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο πάρα πολύ σημαντικά βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας διότι αυτό το οποίο ονομάζεται ευρωπαϊκό χρήμα, δηλαδή η πόρη των ιδιωτικών ταμείων, είναι κάτι το οποίο ετώνωσε την οικονομία μας και κατά τρίτον τώρα ωφελούμεθα από την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων στην Ένωση και τώρα πια έχουμε συνηθίσει στην περιοχή Σέγγεν να διακινούμεθα ελεύθερα οπότε τώρα ελεύθερα μπορούμε να πάμε να σπουδάσουμε, να εργαστούμε, να κερδίσουμε εμπειρίες επισκεπτόμενοι τα άλλα κράτη-μέλη. Κατά τέταρτον, η ελευθερία υπηρεσιών αλλά και εμπορευμάτων είναι κάτι πάρα πολύ βασικό για τις επιχειρήσεις μας. Κάθε επιχειρηματίας, κάθε καταναλωτής τώρα γνωρίζει ελευθερία, την ελευθερία του ότι δεν υπάρχουν φραγμοί τελωνιακοί ή άλλου είδους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την δική μας χώρα, γιατί η δική μας αγορά είναι ιδιαίτερος μικρή. Ε, κατά πέμπτον και ε, πάρα πολύ σημαντικό, η φωνή της χώρας μας τώρα ακούγεται στην Ευρώπη, αλλά ακούγεται ε, και παντού σε όλο τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Φωνή στη συνέχεια, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ότι υπάρχει ένας μηχανισμός συνεργασίας μοναδικός, ο οποίος μας επιτρέπει να μπορούμε να αναζητήσουμε κάποιες δυναμικές, ενεργητικές ε, λύσεις για κάποιες προκλήσεις, κάποια προβλήματα όπως το δημογραφικό, όπως το κλιματολογικό, το ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις βιώσιμες για το ενεργειακό, για το πρόβλημα της μετανάστευσης, αλλά και να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά την χρηματοπιστωτική κρίση. Η Λετωνία βεβαίως και ωφελήθηκε από τα μέσα οικονομικής και οικονομικής πολιτικής. Όμως, αναλάβαμε και τις ευθύνες μας και γίναμε πιο υπεύθυνοι στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Ε, και αυτή την ευθύνη την έχουμε έναντι των Ευρωπαίων, των Ευρωπαϊκών λαών. Επίσης θα πρέπει να ρίξουμε μια μεθιά στα λάθη που έγιναν στο παρελθόν προσχωρήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ο βασικό στόχο ο οποίο επετεύχθη. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, επαναπαυθήκαμε στι ε, δάφνε μα, χωρί να συνειδητοποιήσουμε πλήρω ότι βρισκόμαστε στην αρχή και όχι στο τέλο αυτή τη εξελικτική διαδρομή, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει αν σωρεύει ευκαιρίε, όμω απόκειται σε κάθε κράτο μέλο το πώ θα τι εκμεταλλευτεί. Εμεί δεν εκμεταλλευτήκαμε όλε τι ευκαιρίε που προσφέρθηκαν δεν ε, χρησιμοποίησαμε τα, τα μέσα συνοχής ε, πλήρως ούτε τα χρηματοδοτικά μέσα. Ακόμα μαθαίνουμε, ακόμα οι κυβερνήσεις μας ε, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτές μας τις ευρωπαϊκές επαφές. Βεβαίως χάσαμε και το τρένο του ευρώ, κάτι το οποίο ήταν ένα λάθος, το οποίο τώρα που μας χτυπάει η οικονομική κρίση είναι κάτι το οποίο φαίνεται πολύ. Όμως ακόμα και πιο σκληροί ευρωσκεπτικοί θα πρέπει να σκεφτούν ότι ο απολογισμό είναι θετικό από την ένταξη. Κανένα. στη Λετωνίδα θα ήθελε να γυρίσει τότε που είχαμε τα τελωνιακά σύνορα και φραγμού. Κανεί δεν θέλει να κάνει αυτέ τι τεράστιε ουρές για να μπορέσει να περάσει τα σύνορα, κάποια σύνορα. Ούτε κανεί στη Λετωνία θα ήθελε να ξαναέχουμε ε, φραγμούς και περιορισμούς όσον αφορά την μετακίνηση φοιτητών, σπουδαστών, εργαζομένων. Οπότε βλέπουμε ότι οι ευρωσκεπτικιστές πάβουν να είναι ευρωσκεπτικιστές βλέποντας αυτά όλα τα θετικά. Τώρα έχουμε αυτή την βαθιά κρίση, οπότε η οικονομία έχει υποστεί χτύπημα, η κατάσταση επιδεινώνεται και λίγα μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις, βλέπουμε Μέχρι σήμερα είχαμε ελεύθερη ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και εμείς πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν η αγορά να διέπεται από την αυτορύθμιση θεωρούμε ότι η αγορά είναι κάτι το πάρα πολύ βασικό. Θεωρούμε ότι τα πράγματα θα διορθωθούν. Αυτό ήταν στο παρελθόν κάτι το οποίο πιστεύαμε, όμως είδαμε τι έγινε με αυτή την κρίση, πόσο, πόσο χτυπήθηκε το, η οικονομία μας και το οικονομικό αυτό σύστημα. Και το χειρότερο είναι ότι ο μέσος άνθρωπος ε, χτυπήθηκε πάρα πολύ σοβαρά, Είδαμε τι έγινε κατά τα τέλη του παρελθόντος έτους, κάτι το οποίο επίσης έδειξε το ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν πιο δυναμικό ρόλο στο οικονομικό προτσέ. Θα πρέπει επομένως να κρατάμε το επιτέλεσμα της ε, οικονομίας με υπεύθυνο τρόπο, με επαγρύπνηση. Δυστυχώς ε, συνήλθαμε πάρα πολύ αργά ε, είδαμε ότι το, τοπιδάλιο, πιδάλιο το, το είχαμε αφήσει ανεξέλεγκτο και το πλοίο πήγαινε προς τα βράχια. Θα πρέπει τελευταία στιγμή να αλλάξουν πορεία, να βρούμε μια λύση για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Γιατί όλοι χρειάζονται μια συντονισμένη αντίδραση, λύση για να ξαναμπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης για να μπορέσουμε να εξεύρουμε μηχανισμούς οι οποίοι θα βοηθήσουν το σύστημα, το οικονομικό, να υπάρξει μηχανισμός εποπτείας και ελέγχου, αλλά από την άλλη μεριά να μην επιβάλλουμε κάποιους περιορισμούς όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς. Να βρούμε μια ισόρροπη προσέγγιση, αυτό είναι η σημερινή πρόκληση. Εμείς, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα του ότι μπορούμε να συντονίσουμε τις εθνικές δραστηριότητες. Και έτσι να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο και μια ενιαία λύση. Με μεγάλη μας χαρά διαπιστώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτό το πρόγραμμα ε, <clears throat> για να βοηθήσει την ε, ευρωπαϊκή οικονομία να βγει από την κρίση. Υπάρχουν και εθνικές λύσεις. Η κρίση έπληξε και τη δική μας χώρα. Έχουμε ίσως, ίσως από τις πιο εντυπωσιακέ ε, κρίσεις στη χώρα μας και θα πρέπει να βρεθούν κάποιες, ε, κάποια, κάποια κίνητρα ώστε σύντομα να μπορέσουμε να, να την οικονομία μας ε, κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Όμως η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί. Να έχουμε ξεκάθαρο όραμα, να μην έχουμε κοντόφθαλμες λύσεις κατά νου, αλλά να βλέπουμε πιο μακριά. Κατά τα τέλη του 2008, έξι κυβερνήσεις αλλά και κόμματα της Συγγνώμη, η κυβέρνηση και έξω της συμφώνησαν για ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο ε, πρότεινε η κυβέρνηση. Θα έχουμε τώρα ε, κάποια υποπτία, έλεγχο του τι θα γίνουν τα κρατικά δάνεια. Ε, τάξαμε κάποιες μεσοπρόθεσμες προτεραιότητές μας, ε, διευκόλυνση των εξαγωγών, εγγύηση ε, για έναν αθέμητο δίκαιο ανταγωνισμό, αντιμετώπιση του τρέχοντος χρέους και το 2012 θέσπιση του ευρώ. Η δε είσοδός μας στην Ευρωζώνη έχει καταστεί ένα στρατηγικός μας στόχος. Έτσι θεωρούμε ότι θα πετύχουμε μακροπρόθεσμα την οικονομική σταθερότητα. Ευτυχώς δεν είμαστε μόνοι στην αντιμετώπιση της κρίσης. Όχι μόνο οι διεθνείς φορείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κρατημέλη μας βοηθούν να βγούμε από αυτές τις δύσκολες μέρες και σας ευχαριστούμε για την αλληλεγγύη σας. Κυρίες και κύριοι, με κάθε διεύρυνση, νέες χώρες μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά κάθε φορά άλλαζαν και οι προτεραιότητες. Εμείς όταν μπήκαμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε ω καινούργια πολιτική πολιτική γειτονία. Οπότε και είχαμε και ένα σωρό μέσα πολιτική, εφαρμοστικέ διατάξει και έτσι ε, άλλαξε η πολιτική προς τα ανατολικά σύνορα της ε, Ευρώπης. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με τα νέα κράτη-μέλη. Εμείς πάντα βλέπουμε όσο γίνεται πιο πλατιά αυτήν την πολιτική γειτονίαση και προσπαθούμε με ενεργά να βοηθήσουμε στην υλοποίηση αυτή τη πολιτική. Γιατί δεν πρόκειται εδώ μόνο για τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και των γειτόνων τη. Όσον αφορά δηλαδή τα χερσαία και θαλάσσια σύνορα τη Ένωση. Στα πλαίσια τη πολιτική γενίαση. θα πρέπει να δούμε τον ρόλο της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα. Εμείς ανέκαθεν θεωρήσαμε ότι θα πρέπει προς Ανατολάς να είναι πιο ενεργή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και είχαμε διάφορες πρωτοβουλίες, εταιρικέ σχέσεις, ούτω ώστε να λάβουμε υπόψη, να λάβουμε υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ιδιορυθμίες αυτής της περιοχής της Ευρώπης. Οπότε είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική φιλόδοξη. Γι' αυτό και χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες της σχετικής ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι εταιρικές σχέσεις προς Ανατολάς θα ε, κάνουν πιο στενές τις οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τους προσανατολάς γείτονες. Επίσης θα έχουμε πιο στενή συνεργασία. Θα πρέπει να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία. Να προσέξουμε το ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση κατά περίπτωση να αξιολογούμε ε, το, το κάθε κράτος χωριστά και να δούμε ξανά τους στόχους μας που θα τους πετύχουμε μόνο εάν συνεργαστούμε με όλες τις χώρες αυτής της περιοχής. Να βοηθάμε όποτε όποιον το χρειάζεται. Επίσης, ήταν πάρα πολύ θετική η υποδοχή της πρότασής μας για περισσότερη συνεργασία στις χώρες Κεντρικής Ασίας, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν. Εμείς ανέκαθεν ήμασταν υπέρ του να εφαρμοστεί η πολιτική γειτονία και για εκείνες τις χώρες. Αυτό το πιστεύαμε και θα συνεχίσουμε να το πρεσβεύουμε και έτσι θα βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις μας. Η κάθε μία από αυτές τις χώρες έχει κάποια ιστορική εμπειρία, όλοι μπορούν να συμβάλλουν σε μια κοινή πορεία. Εμείς βοηθούμε επομένω όσον αφορά αυτή την ε, πτυχή της προσανατολάς πολιτική και ε, έχουμε γνώσεις ιστορικές αυτής της περιοχής της Ευρώπης. Θέλουμε επομένω να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γνώση, να την εφαρμόσουμε, να μην πάει χαμένη, ε, να μην χάσουμε το τρένο τη εκμετάλλευση των ευκαιριών για την επόμενη δεκαετία. Δεν θέλουμε η Λετωνία να είναι ακόμα μία χώρα για τι προσανατολέ χώρε. Θέλουμε η Λετωνία να είναι μία πύλη προ την Ευρώπη. Και έτσι ε, θέλουμε να συνεχίζεται ένα ε, ενεργητικό, δυναμικό, διάλογο και οι γειτονέ μα να καταλάβουν καλύτερα τι ευρωπαϊκέ αξίε να καταλάβουν ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και οι στόχοι της προσανατολάς εταιρικής σχέσης και με αυτή την ευκαιρία και εμείς βέβαια να αφουγκραστούμε τους γείτονες, να μάθουμε τι όραμα έχουν για το μέλλον, τι σχέση θέλουν να έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θεωρούμε ότι θα είναι κέρδος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και γι' αυτό και θέλουμε να υπάρχει ιδιαίτερη ε, πρόθεση τη εταιρική σχέση προσανατολά κατά την τσεχική προεδρία. Κατά τι πρώτε ημέρε, οποίε είχαμε βέβαια όπως ξέρετε, ε, την ανάδειξη της ενεργειακής πολιτικής ως κάποιο θέματο πολύ σημαντικού. Γιατί χρειάζεται να βρούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να φτάσουμε σε ενεργειακή ασφάλεια. Αυτό, επομένως, θα είναι ένα θέμα πάγιας ε, και υψηλής προτεραιότητας. Είναι κάτι που θα μας απασχολεί περισσότερο κάθε μέρα. Η ενεργειακή ασφάλεια έχει και μια εξωτερική διάσταση πάρα πολύ σημαντική. Ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε το ενεργειακό απομονωμένα από τις πρόσφατες εξελίξεις. Είδατε τι έγινε στη Γεωργία αλλά και στην Ουκρανία γιατί ακόμα και στο πρόσφατο παρελθόν ε, τα κράτη-μέλη θεωρούσαν ότι είναι εθνικό θέμα το ενεργειακό και όχι κάτι πρέπει να το μετωπιστεί σε ενωσιακό επίπεδο. Είδαμε όμως τα τελευταία χρόνια τι έγινε. τι έγινε με, το, με τις ενδιακές πηγές, ε, με τις διακοπές στην προμήθεια. Άρα χρειάζεται να υπάρξει μια ενιαία ενεργειακή πολιτική. Όπως έχει σήμερα η κατάσταση, ο βασικός πολιτικός στόχος είναι να έχουμε τακτή, επαρκή, βιώσιμη αλλά και περιβαλλοντικά σωστή ενεργειακή πολιτική. Είναι αλήθεια ότι ήταν κάπως άνηση η πορεία μας σε αυτά τα θέματα. Άρα χρειάζεται ενεργειακός τομέας πράσινος. Είναι φιλόδοξοι στόχοι που έχουμε τάξει, θα πρέπει να τους πετύχουμε όμως. Και βρισκόμαστε νομίζω μόνο στην αρχή μιας μακράς πορείας όσον αφορά το να έχουμε περισσότερες εναλλακτικές όσον αφορά την προμήθεια ενέργειας. Η διακοπή της παροχής από την Ρωσία είναι κάτι που μας άνοιξε τα μάτια. Είδαμε ότι χρειάζεται ταχύως να εξευρεθεί λύσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είναι δική μα ευθύνη. Επομένω, αυτή η κοινή κατανόηση του προβλήματο θα πρέπει να υλοποιηθεί στην ε, κατοχήρωσή μα στο να έχουμε περισσότερες, ε, περισσότερες πηγές ενέργειας να μην λιώσει σαν το χιόνι την άνοιξη αυτή μας η συνειδητοποίηση ε, τόσο ο προβληματισμός να γίνει ένας διάλογος διάλογος δυναμικός με τις χώρες που μας παρέχουν την ενέργεια και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Έχουμε δε ως όπλα ε, τις πολιτικές μας. Ολοκλήρωσε επίσης να υπάρξει στην ενεργειακή ε, αγορά ε, όσον αφορά την περιοχή της Βαλτικής, Γερμανίας και Σκανδιναβίας. Εκεί επίσης είχαμε κατάσταση και εξέλιξη άνηση, είχαμε και κάποιες περιόδους στασιμότητας. Βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλά προσπάθησε να εξασφαλίσει ελληνική και πάρκια για την Ευρώπη. Γι' αυτό και είχαμε αυτό το δίκτυο ε, και διασύνδεση των βαλτικών αγορών. Τελικά θέλουμε να μπει στην κοινή ενεργειακή αγορά όλη η Βαλτική. Πάρα πολύ θετικό ήταν το πόσο βοήθησε σε αυτές τις στρατηγικές προσπάθειες η Σουηδία, η οποία θα έχει ευκαιρία ε, κατά το δεύτερο εξάμεινο, κατά την προεδρία της, φέτος να δουλέψει περισσότερο αυτό το ζήτημα και είμαστε ε, πεπισμένοι ότι ισχυρές περιφέρειες σημαίνουν ισχυρή Ευρώπη και αυτό αφορά και τη Βαλτική θάλασσα αλλά και τη Μεσόγειο θάλασσα. Κυρίε και κύριοι, το ευρωπαϊκό όραμα ήθελε ανέκαθεν να, να πετύχει ευημερία για τους Ευρωπαίους. Τώρα όμως κάποια πράγματα έχουν αλλάξει, έχουμε τώρα παγκοσμιοποίηση, διασύνδεση πολύ περισσότερο των οικονομιών ανά τον κόσμο από ό,τι πριν μια πεντηκονταετία. Έχουμε νέους παίκτες, νέους πρωταγωνιστές στην σκηνή και μόνο εάν ε, έχουμε μακροπρόθεσμο όραμα, αν είμαστε ενωμένοι, αν είμαστε συνεπείς, τότε μόνο θα βγούμε χαμένοι από αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι του ανταγωνισμού. Μόνο χέρι-χέρι, αν προχωρήσουμε, θα πετύχουμε την ευημερία που θέλουμε και θα πετύχουμε τους στόχους τους οποίους τάξαμε και για τους οποίους μας εξέλεξαν οι λαοί. Επανειλημμένα απέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι μπορεί να προσφέρει μια προοπτική ευρύτερη για το μέλλον της Ευρώπης. Πάντοτε έχει ισόρροπη και δίκαιη προσέγγιση στο θέμα της ε, διεύρυνσης. Έτσι η Ευρώπη έγινε πιο ανταγωνιστική, έτσι γνώρισε η Ευρώπη κάποια ανάπτυξη. Αυτά όλα είναι όπλα, ατού πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε και για τη Λατινική Αμερική και για την Ασία είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πρωταγωνιστής η Ευρώπη. Εσείς ξέρετε τι ευθύνε έχουμε για όλη αυτή τη διαδικασία και βεβαίως και ξέρουμε πόσο εσείς μπορείτε να φέρετε το ευρωπαϊκό όραμα κοντά στους Ευρωπαίους. Στο μέλλον θα πρέπει να έχετε πιο σημαντικές αρμοδιότητες, θα πρέπει να υλοποιήσετε την ενότητα στην διαφορετικότητα ως ιδέα και θα πρέπει σε συνεργασία να προχωρήσουμε για τους κοινούς στόχους που είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλά είναι επίσης σημαντικό να μην έχουμε πολυδιάσπαση στην Ευρώπη θα πρέπει να βρίσκουμε κάποιες λύσεις και ίσως να μπορέσουμε να καταφέρουμε μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Έχουμε τη συνέχεια της Λισαβόνας, έχουμε την σχετική συμφωνία του περσμένου μήνα και θεωρούμε ότι αυτή η συνθήκη είναι προϋπόθεση εύρεθμης λειτουργίας της Ευρώπης, προϋπόθεση για ενίσχυση της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή. Και μόνο εάν υλοποιήσουμε τις αρχές της Λισαβόνας, τότε μόνο θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες μας τις δυνατότητες, Δυνατότητε μια μιας ενωμένης νέας Ευρώπης. Όμως, στην πράξη, το πώς θα πιάσει από αυτή η συνθήκη θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση κρατών, θεσμικών οργάνων και από τη δυνατότητά μας να είμαστε ενωμένοι και αλληλέγγυοι, κυρίε και κύριοι. Μέχρι το 2004 θέλαμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε οι στόχοι μας είναι οι στόχοι όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν αποτελούμε ένα απόσπαστο τμήμα της Ευρώπη. Η Λετωνία έχει τους στόχους αυτούς που ταιριάζουν με το ευρωπαϊκό όραμα. Και είναι δεδομένο να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και τους θέλουν όλα τα κράτη-μέλη. Θεμέλιο είναι οι κοινέ αξίε, αυτό το θεμέλιο τη Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί. Όσον αφορά δε τις ε, κοινέ αξίες είναι αυτές οι οποίες ε, βοηθούν το να γίνεται διάλογος για όλα τα ζητήματα και αυτά ακριβώς αποτελούν το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο στόχος όλων των πολιτικών και όλων των ηγετών της Ευρώπης να ενθαρρύνουν ε, τον προβληματισμό για αυτές τις κοινέ αξίες για το μέλλον τώρα. Πώς βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς βλέπουμε την Λετωνία το 2015. Καταρχήν Θεωρούμε ότι θα υπάρχουν διάφορα κέντρα αποφάσεων που θα έχουν διαμορφωθεί μετά την οικονομική κρίση. Ένα από τα κέντρα αυτά θα είναι η Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να μπορέσει να είναι ενωμένη, γιατί μόνο με την ενότητα μπορούμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Επίσης, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε όλους τους Ευρωπαίους οι οποίοι ασπάζονται τις κοινέ αξίες. Ενότητα στη διαφορετικότητα, αυτό είναι το κλειδί για την εξασφάλιση του μέλλοντος. Διεύρυνση της Ευρώπης, αλλά και διατήρηση της αποτελεσματικότητας. Θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να έχει κάποια πολιτική ασφάλειας, κάποια πολιτική σταθερότητας και σε σχέση με τους γείτονες. Στα πολιτιστικά, στα θέματα της παιδείας, ε, εκεί θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την πολυμορφία, τον πλούτο των διαφορετικών ε, παραδόσεων και να μην έχουμε διαχωρισμό μεταξύ μικρών, μεγάλων, παλιών και καινούργιων κρατών μελών. Θα πρέπει ο καθένας να κρίνεται όχι γεωγραφικά, όχι γεωπολιτικά, αλλά επί τη βάση των επιδόσεων και επιτευγμάτων του. Ενότητα, ισχυρές περιφέρειες, στενή συνεργασία. Έτσι, όλοι θα βοηθήσουν όσον αφορά την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ευρώπη ο καθένας, αν δούμε τις δυνατότητες, με τις γνώσεις του, μπορεί να βάλει το λιθαράκι του. 2015, ποιος θα είναι ο δικός μας ρόλος τώρα. Η Λετωνία και η Ρήγα μετά την κρίση θα αποτελεί οικονομικό κέντρο για την Βαλτική περιοχή. Θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Θα έχουμε διαρθρωτικά αλλάξει πάρα πολύ. Το 2015 για πρώτη φορά ή στην ιστορία μας ως κρατήτου κράτους θα μπορέσουμε να αναλάβουμε το πιδάλιο της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Έτσι θα βοηθήσουμε. Θα βοηθήσουμε γιατί έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τους γείτονες προς Ανατολάς. Θα είμαστε μία γέφυρα της Ένωσης προς Ανατολάς, όπως έχει συμβεί και με τις χώρες της Μεσογείου προς Νότον. Έτσι θα βοηθήσουμε το ανοιχτό πνεύμα που έχει η Ευρώπη. Το 2015 δεν απέχει πολύ. Μόλις μία εξαετία κύριε και κύριοι. Μόλις πριν από έναν αιώνα ε, κάποιος ε, μεγάλος ποιητής μας είχε πει ότι οι, οι αλλαγές είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό γιατί που τονώνει τις εξελίξεις και αυτό ισχύει και έγινε όσον αφορά το σύστημα αξιών μας. Ε, είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρώπη. Ενότητα στην διαφορετικότητα, αυτές οι εξελίξεις ε, είναι σημαντικές και επομένως η Ευρώπη του μέλλοντος θα ετράζεται σε αυτήν την αξία. Κυρίες και κύριοι, το πόσο ε, πάει καλά η Ευρώπη αυτό είναι η αποτίμηση των επιδόσεών μας. Και παρακαλώ όλοι οι ευρωβουλευτές να προσπαθήσουν να κατανοήσουν το πόσο ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους το να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό είναι η καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του έργου μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία κατά αυτή την κοινωνική θητεία. Σας εύχομαι Καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή επιτυχία στις ε, ευρωεκλογές. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το λόγο που μας απευθύνατε, για το φιλοευρωπαϊκό σας πνεύμα, για τη στράτευση υπέρ της Ευρώπης. Ακούσαμε από τα χείλη σας που τίμησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που επιβεβαιώνουν αυτό στο οποίο και εγώ πιστεύω, ότι κατά τη διαπραγματεύση για την διεύρυνση στο δεύτερο ήμιση της δεκαετίας του 90 η Λετωνία, η Λιθουανία η Σλοβακία είχαν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εκείνο το οποίο επέμεινε έτσι ώστε η Λιθουανία, η Λετωνία και η Σλοβακία να ενσωματωθούν στις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση. Και με χαρά είδαμε την 1η Μαΐου του 2004 και την συμμετοχή της Λετωνίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε στο θέμα της διεύρυνσης, της ενέργειας. Θα επανέλθω κι εγώ για να απαντήσω σύντομα στι παρατηρήσει σας. Έχουμε βέβαια έναν πολύ υπεύθυνο επίτροπο συμπατριώτη σα, τον κύριο Πίπαλ, ο οποίο την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και τώρα ακόμα στα προβλήματα και την κρίση για το φυσικό αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά ιδιαίτερα σχέση με τη Ρωσία, απέδειξε την ικανότητά του. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πίπαλ σε ενώπιόν σα, κύριε Πρόεδρο τη Λετωνία, για την, ε, για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Και κλείνοντα θα παρατηρήσω το εξή, κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι μαθαίνετε, διδάσκεστε και εσείς κύριε Τονία. Σωστό αυτό. Όμως και εκείνοι ακόμη που βρίσκονται από την αρχή, από τις απαρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διδάσκονται από εσά, από τη δική σας ιστορική εμπειρία. Όταν είμαστε λοιπόν διατεθειμένοι ο ένας να εισακούσει τον άλλον, ο ένας να διδαχθεί από τον άλλον, εμπλουτιζόμεθα και ημέν και είδε. Κερδίζουμε και ημέν και είδε και είμαστε ισχυροί, είμαστε δημοκρατικοί, είμαστε ελεύθεροι όλοι επειδή είμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Λετωνίας. Αγαπητοί συναδελφοί, θα ολοκληρώσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου και προχωρούμε τώρα στην έκθεση.